τροπή. Παραπέμπεται, με συγχωρείτε. Τώρα, έχουμε τις δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής ως προς την έκθεση προόδου της Αλβανίας για το 2012. Δίνω το λόγο στην Υπουργό, στην κυρία Μαρκουλή. Έχετε το λόγο. Uh, thank you, Madam President, uh, honorable members. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρίε και κύριοι βουλευτέ. Χαίρομαι που μπορώ να λάβω μέρο σε αυτή τη συζήτηση απόψε. Η Αλβανία είναι μια σημαντική χώρα στην ε, περιοχή. Συνεργαζόμαστε ευρέω ε, σε πολλού τομεί ε, και έχουμε εκτεταμένο πολιτικό διάλογο. Οι σχέσεις μας είναι όλο και πιο σημαντικές και αντικατοπτρίζουν τη σημασία της Αλβανίας στην περιοχή. Ε, έχουμε κάποιες περιφερειακές πρωτοβουλίες όπως το Περιφερειακό ε, Συμβούλιο Συνεργασία και η διαδικασία την Νοτιοανατολικής Ευρώπη επιπλέον η Αλβανία προείδευσε στο Συμβούλιο Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης το 2012. Θα ήθελα να ευχαριστήσω το Κοινοβούλιο για την συνεισφορά του σε αυτή τη συζήτηση και ειδικά να εκφράσω την εκτίμησή μου στον εισηγητή τον κύριο Χουντή για την ε, δουλειά που έκανε. Νομίζω πως υπάρχουν τα πράγματα στα οποία μπορούν να συμφωνήσουν Συμβούλιο και Κοινοβούλιο. Στα συμπεράσματα που υιοθετήθηκαν χτες το βράδυ, το Συμβούλιο καλωσόρισε την πρόοδο της Αλβανίας για την επίτευξη των 12 προτεραιοτήτων που αναφερθεί στην ε, νομοδότηση της Κομισιόν το 2010. Ο διάλογος με την ε, Κομισιόν έχει βελτιωθεί σημαντικά και έτσι ανοίγει ο δρόμος για να εκπληρωθούν τα πολιτικά κριτήρια για την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Αλβανία εκπληρώνει τέσσερις προτεραιότητες κλειδιά και σύντομα θα εκπληρώσει άλλες δύο. Αυτές αφορούν τη λειτουργία του Κοινοβουλίου, μεταρρύθμιση του εκλογικού νόμου και τη δημόσια διοίκηση. Πρόοδος επίσης έχει συνδυαθεί σε άλλους τομείς που είναι τομείς προτεραιότητας. παραδείγματο χάρη η άρση ασυλίας υψηλόβαθμων ε, αξιωματούχων ε, και δικαστών και επίσης ε, αύξηση της δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων που προέρχονται από έγκλημα το Συμβούλιο. Επίσης σημειώνει την πρόθεση να καταστεί η Αλβανία υποψήφια χώρα αρκεί να συμπληρωθούν οι βασικές μεταρρυθμίσεις ε, στον τομέα της δικαιοσύνης και της δημοσίας διοίκησης και βεβαίω ε, και η αναθεώρηση του κανονισμού του Κοινοβουλίου. Η Κομισιόν στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να αναφέρει αμέσως μόλις σημειωθεί κάποια πρόοδος, λαμβάνοντας επίσης υπόψη το εάν έχει υπάρξει πρόοδος στην καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος. Υπάρχουν και άλλοι τομείς ε, όπου θέλουμε να δούμε περισσότερες προσπάθειες από την Αλβανία. Αυτά είναι ζητήματα κράτους δικαίου, ενίσχυσης της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης, της αποτελεσματικότητας, της ε, λογοδοσίας και τα θέματα μειονοτήτων. Όλα θα είναι υποχρεώσεις προς την Ευρωπαϊκή Ένωση κύριε Πρόεδρε. Κυρίε και κύριοι βουλευτέ, θα ήθελα τώρα να αναφερθώ στι βουλευτικέ εκλογέ του επόμενου έτου. Γνωρίζουμε πω ε, ήταν ε, συχνά αντικείμενο διαφωνιών οι εκλογέ στην Αλβανία. Οι εκλογέ του Ιουνίου θα αποτελέσουν μια ευκαιρία για να επιδείξουν όλα τα πολιτικά κόμματα της Αλβανίας τη δέσμευσή τους στην μεταρρύθμιση της εκλογικής διαδικασίας και ένα σημαντικό τεστ για την λειτουργία της δημοκρατίας και των δημοκρατικών θεσμών. Και επίσης ο πολιτικός διάλογος σε όλους τους τομείς που καλύπτονται από τις ε, προτεραιότητες είναι κρίσιμη σημασία για την πρόοδο της Αλβανίας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ε, Ευχαριστούμε την Υπουργό. Το λόγο έχει ο Επίτροπος Φιούλε. Thank θα ήθελα να ευχαριστήσω το Κοινοβούλιο και δι τον εισηγητή τον κύριο Χουντή για την έκθεση για την Αλβανία. Χαίρομαι που υποστηρίζετε τις ευρωπαϊκές προοπτικές της Αλβανίας και για το ότι αναγνωρίζετε τις δυνατότητες της διαδικασίας ένταξης ως αποτέλεσμα πολιτικής συνεργασίας εντός της χώρας. Η έκθεση ευθυραμίζεται και με τις συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πλαίσιο των, δέσμη της δέσμης για την διεύρυνση. Αφενός με να γνωρίζουμε τα επιτεύγματα της Αλβανίας, αφετέρου δε τονίζουμε την σημασία να συνεχιστούν οι μεταρρυθμίσεις στην Αλβανία σε όλους τους τομείς στο πλαίσιο των 12 προτεραιοτήτων που εντοπίζει η Κομισιόν στην γνώμη της του 2010 εν ώψη της αίτησης της Αλβανίας να γίνει μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η έκθεση του 2012 της Κομισιόν έχει νέα ευρήματα. Αντικατοπτρίζει τη νέα κατάσταση στην χώρα. Καταγράφει την πολιτική συμφωνία του Νοεμβρίου του 2011 μεταξύ της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης. Συμφωνία με την οποία τερματίζεται η τελμάτωση τη πολιτική κατάσταση και εγγενιάζεται περίοδο συνεργασία μεταξύ των πολιτικών δυνάμεων, κάτι το οποίο κατέστησε και τι δυνατέ τη μεταρρυθμίσει βάσει των προτεραιοτήτων που είχε αναδείξει η Κομισιόν. Με βάση αυτήν την πρόοδο, η Κομισιόν προτείνει να χορηγηθεί το καθεστώ τη υποψηφία χώρα στην Αλβανία με την προπόθεση βελτιώσεων στην δικαιοσύνη και στην δημόσια δίκηση καθώς και όσον αφορά την τροποποίηση των κανόνων λειτουργίας του Κοινοβουλίου. Η Αλβανία πρέπει να συνεχίσει να προβαίνει σε μεταρρυθμίσεις. Δυστυχώς οι πολιτικοί ηγέτες της χώρας δεν μπόρεσαν σε όλες τις περιπτώσεις ε, να ανταποκριθούν στι απαιτήσει αυτέ με τρόπο συνεπή. Ούτε ήταν η προτεραιότητα αυτή πρώτη προτεραιότητα για την αλβανική κυβέρνηση δεν κατάφεραν να πετύχουν και τους απαραίτητους πολιτικούς συμβασμούς για να προβούν δηλαδή σε ριζικές μεταρρυθμίσεις. Οι προποθέσει βεβαίω υπάρχουν, γι' αυτό πρέπει να συνεχίσουμε να ενθαρρύνουμε του Αλβανού φίλου και την κυβέρνηση αλλά και την αντιπολίτευση να εστιάσουν τη δράση του στην διαδικασία ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πέρα από τα βραχυπρόθεσμα μέτρα τα οποία προανέφερα, η Αλβανία αντιμετωπίζει πολλές προκλήσεις και ιδιαίτερα στον τομέα του κράτους δικαίου και το οποίο υπογραμμίζετε κι στο ψήφισμα. Αυτό εννοείται ότι απασχολεί και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρέπει να ενστερνιστεί η πολιτική τάξη της αλλαγή. Αυτό είναι κάτι απολύτως απαραίτητο. Η Αλβανία θα χρειαστεί να αξιοποιήσει τα ήδη σημειωθέντα επιτεύγματα, θα πρέπει να τα παγιώσει και να συνεχίσει σε βιώσιμη βάση τον πολιτικό διάλογο. Όλα αυτά είναι προαπαιτούμενα για να μπορέσουν να έχουν απόδοση και αποτέλεσμα οι μεταρρυθμίσει. Επίση, πρέπει η Αλβανία να αποδείξει ότι μπορεί να πετύχει περισσότερα στον αγώνα κατά τη διαφθορά, του ξεπλήματο του οικονομικού χρήματο και κατά του οργανωμένου εγκλήματο. Η επιτυχής διεξαγωγή των εκλογών τον Ιούνιο του 2013 θα αποδείξει για άλλη μια φορά τις ευρωπαϊκές προοπτικές της Αλβανία. Συμμεριζόμαστε τη γνώμη σα όσον αφορά τι καλέ σχέσει γειτονία και τη συμβολή τη Αλβανία στην σταθερότητα τη περιοχή. Και αυτά είναι προαπαιτούμενα για την συνέχιση περαιτέρω τη διαδικασία ένταξη. Πρέπει να στείλουμε ένα στεναρό μήνυμα προ την Αλβανία και να την καλέσουμε να συνεχίσει τι επικοδομητικέ της προσπάθειε στην περιοχή υπογραμμίζοντα προ του πολιτικού τη ηγέτε, την σημασία των σαφών πολιτικών μηνυμάτων, των καλών πολιτικών σχέσεων και των καλών σχέσεων γειτονία. Ευχαριστώ πολύ για άλλη μια φορά, κυρίε και κύριοι βουλευτέ, για την υποστήριξή σα, απαραίτητη για την συνέχιση της διαδικασίας διεύρυνσης. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Εξ ονόματος τώρα των πολιτικών ομάδων αρχίζοντας από τους σοσιαλιστές, όχι με συγχωρείτε λέει η Πρόεδρος, από την ΚΟΕ έχει το λόγο ο κύριος Χουντής για δύο λεπτά. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, παρά το γεγονός ότι η έκθεσή μας, η έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την ενταξιακή προοπτική της Αλβανίας συζητείται σχεδόν ταυτόχρονα με το Συμβούλιο, το οποίο παίρνει και τις αποφάσεις, τις αποφάσεις τις οποίες μας ανέφερε η κυρία Υπουργός, νομίζω ότι η έκθεση του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου έχει τη σημασία της. η έκθεση υπερψηφίστηκε από την επιτροπή εξωτερικών υποθέσεων από όλες τις πολιτικές ομάδες γι' αυτό θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους ιδιαίτερα τους σκιώδεις συζητητές, για την συμβολή και τη στήριξή τους. αγαπητοί συνάδελφοι η έκθεση για την ενταξιακή προοπτική της αλβανίας για άλλη μια φορά υπογραμμίζει το γεγονός ότι εφόσον η ένταξη της αλβανίας στην ευρωπαϊκή ένωση είναι επιθυμία του αλβανικού λαού εμείς οφείλουμε αυτή την επιθυμία να τη σεβαστούμε και να δημιουργηθεί το κίνητρο για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που έχει προβλήματα δημοκρατίας προβλήματα κράτους δικαίου να χτυπηθεί διαφθορά να λυθούν μειωνοτικά εργασιακά δικαιώματα. με αυτή την έννοια η υπόθεση της ένταξης είναι υπόθεση της αλβανικής κοινωνίας όχι απλώς των αλβανικών δυνάμεων. θέλω να πω λοιπόν ότι έχουν γίνει βήματα πρέπει να γίνουν ακόμα περισσότερα η έκθεση επισημαίνει ορισμένα από αυτά. όμω κύριε επίτροπε και κυρία υπουργέ θα ήθελα να σταθώ στι πρόσφατε δηλώσει του αλβανού πρωθυπουργού. δηλώσει έγιναν μετά την επιτροπή που ενέκρινε το ψήφισμα που δημιούργησαν ένταση και υπονόμευσαν το κλίμα και τι σχέσει καλή γειτονία στην περιοχή. παρά την προσπάθεια να ανασκευαστούν νομίζω ότι πρέπει τέτοιε τοποθετήσει και αντίστοιχε πρακτικέ εθνικιστικού και αλυτρωτικού περιεχομένου και να αποφεύγονται δεν δικαιολογούνται κάτω από οποιαδήποτε σκοπιμότητα αφορούν μια πολύ ευαίσθητη και πολύ πάθη περιοχή όπω τα βαλκάνια. με αυτή την έννοια αγαπητοί συνάδελφοι το ευρωπαϊκό κοινοβούλιο και οι άλλοι ευρωπαϊκοί θεσμοί θα πρέπει να σταθούν αυστηρά και αποφασιστικά σε τέτοιε αντιλήψει ούτω ώστε και να απαιτήσουν να ενισχυθούν οι σχέσει καλή γειτονία τη αλβανία με τι άλλε χώρε όχι μόνο για να κρατηθεί ζωντανή η ενταξιακή προοπτική της αλβανίας αλλά για την ασφάλεια τη σταθερότητα και την ειρήνη στην περιοχή. σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Εκ μέρους του ΕΛΚ, ο κύριος Κούκαν, για δύο λεπτά. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Χαιρετίζουμε την έκθεση αυτή και θα θέλαμε να συγχαρούμε και τον εισηγητή. Συγχαρητήρια και τους, τους ε, Αλβανούς για τα επιτεύγματά τους. Θα θέλαμε να τους ενθαρρύνουμε να ποντάρουν πάνω σε αυτό. Η Επιτροπή μας έστειλε, ένα θετικό μήνυμα στην ε, Αλβανία συστήνοντας να αποκτήσει καθεστώς υποψήφιας χώρας υπό τον ορό ότι θα πληρωθούν οι οκτώ προϋποθέσεις. Πιστεύουμε ότι αυτό θα πρέπει να αποτελέσει κινητήριο δύναμη για την Αλβανία κατά τη διάρκεια της ένταξης στην Ευρώπη. Και πιστεύουμε ότι αυτό είναι καθοριστικής σημασίας για τους παρακάτω λόγους. Καταρχάς, το χρονοδιάγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν θα πρέπει να αποτελέσει ένα αντικείμενο διαπραγμάτευσης εσωτερικής πολιτικής. Θα πρέπει να είναι ένας ενοπητικός παράγοντας. Η έκθεση εκφράζει την εκτίμησή της για τις προσπάθειες που έχουν καταβληθεί. Θα πρέπει όμως να αναφέρουμε ότι ο πολιτικός διάλογος και η πολιτική συνεργασία δεν μπορεί να είναι επιλεκτικές. Θα πρέπει να βασίζονται να είναι δρεωμένα μέσα στο σύστημα. Βεβαίως υπάρχουν ορισμένες ανησυχίες σε ό,τι αφορά αυτό το θέμα. Δεύτερον, ναι, η Ευρωπαϊκή Ένωση υπήρξε απόλυτα σαφής ως προς τα προσδοκόμενα από την Αλβανία. Θα πρέπει να υπάρξουν προτεραιότητες ή να περάσουν με στα επόμενα βήματα. Η αξιοπιστία της διαδικασία θα πρέπει να βασίζεται σε ορισμένες προϋποθέσεις και θα πρέπει να γίνουν σεβαστά όσα συμφωνήθηκαν. Τέλος, η Αλβανία έχει πιθανότητες στο μέλλον να, να εντεθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση Έχουμε μια ιδιαίτερα ενθαρρυντική έκθεση. Είναι οι εκλογές αποτελούν μια μεγάλη ευκαιρία για να δείξει η Αλβανία πόσο υπάρχουν μηχανισμοί και πολιτικοί που έχουν βαθιές ρίζες στις δημοκρατικές αξίες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Για την ομάδα σοσιαλιστών και δημοκρατών ο συνάδελφος Ρούτσακ. Ευχαριστώ το κύριε Πρόεδρε, κύριε Πίτρο, αγαπητοί συνάδελφοι. Η ομάδα μου, η ομάδα των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών θα επιθυμούσε να υποστηρίξει την ένταξη της Αλβανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σήμερα συζητήσαμε την έκθεση πρόοδου η Αλβανία τους τελευταίους 12 μήνες επιτέλεσε σημαντική πρόοδο. Η πρόοδος αυτή βασίζεται στη συνεργασία μεταξύ των βασικών πολιτικών δυνάμεων στην Αλβανία. Δίχως αυτή τη συνεργασία μεταξύ της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης δεν θα είχε καταστεί δυνατή η επίτευξη αυτής πρόοδου. Θα ήθελα λοιπόν να απευθυνθώ στους Αλβανούς φίλους και στην κυβέρνηση και στην αντιπολίτευση να συνεχίσουν έτσι. Γιατί δίχως αυτή τη συνεργασία δεν θα μπορέσει να επιτευχθεί περαιτέρω πρόοδος στους τομείς αυτούς που ανέφερε και ο υπουργό και ο Επίτροπος. Αυτό που θα είναι καθοριστική σημασία του χρόνου θα είναι οι εκλογές, όχι το, απο, το αποτέλεσμα, η εκλογική διαδικασία πριν και μετά τις εκλογές. Στις τελευταίες εκλογές, ε, τις βουλευτικές και τις περιφερειακές, ε, ανέκυψαν πολλά προβλήματα. Είναι σημαντικό τον Ιούνιο του 2013 αυτή τη φορά να, να καταγραφεί μία πρόοδο σε ό,τι αφορά τη διεξαγωγή θα ήθελα να αναφερθώ σε ένα θέμα, το θέμα της περιφερειακής συνεργασίας. Μέχρι τώρα η Αλβανία διαδραμάτισε ιδιαίτερα θετικό, ιδιαίτερα επικοδομητικό ρόλο σε ό,τι αφορά την περιφέρεια, σε ό,τι αφορά την, το κοσυφοπαίδιο, το, φύ, το Ο κύριος Χουντής ανέφερε ότι πρόσφατα υπήρξαν ε, υπήρξε ένα δικηστικό κείμενο στα ε, τύρανα. Δεν νομίζουμε ότι είναι σωστό αυτό για την Αλβανία ούτε για την περιφέρεια. Θα θέλαμε λοιπόν να ζητήσουμε από την κυβέρνηση και από την ε, αντιπολίτευση να αποφύγουν αυτού του είδου την ρητορική. Η Αλβανία παίζει καθοριστικό ρόλο για μας. Είναι μια πολύ σημαντική ε, ε, χώρα. Ο ρόλος που διαδραμάτισε ήταν ιδιαίτερα επικοδομητικός και ελπίζουμε να συνεχίσει την ίδια τραπό κινούμενοι προς την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει η συνάδελφος Κορνέλισεν για 1,5 λεπτό για την ομάδα των Πρασίνων. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Μια από τις κύριες ανησυχίες μας σε σχέση με την Αλβανία είναι πάντα το πολιτικό κλίμα. Η απουσία βούλησης για συνεργασία μεταξύ των κυρίων παραγόντων στη χώρα και των κυρίων κομμάτων. Φαίνεται ότι αυτό έχει κάπως αντιμετωπιστεί, είχε μάλλον αντιμετωπιστεί στο παρελθόν και είχε αρχίσει να λειτουργεί ικανοποιητικά σχετικά το κοινοβούλιο. Τώρα όμως δυστυχώς δεν είμαστε τόσο ε, σίγουροι ότι αυτό ισχύει. Πέρασαν τρεις διαφορετικές προτάσεις ε, μέσα σε μια ε, ανεξέλεγκτη κατάσταση αντιπαραθέσεων. Ο Πρωθυπουργό Μπερίσα ανακοίνωσε ότι μπορεί να χορηγήσει αλβανικό διαβατήριο σε Ανθρώπου Αλβανική καταγωγή. ξέροντα τι σημαίνει αυτό για την ευρύτερη περιφέρεια και καθώ είναι και έμπειρος πολιτικός, διερωτώμεθα γιατί το πράττει. Μια επίσκεψη που είχε προβλεφθεί για την προσεχή εβδομάδα, θα ήμουν και εγώ μεταξύ αυτών, αναβλήθηκε τελευταία στιγμή, ματαιώθηκε καλύτερα. Εγώ σκοπεύω να πάω και περίμενα να έχω και επικοδομητικό διάλογο και με την κυβέρνηση και με την αντιπολίτευση. Αλλά από ό,τι φαίνεται οι δεν ήταν διατεθειμένοι να το πράξουν και διερωτώ γιατί. Όλα αυτά πριν από μια πολύ σημαντική συνεδρίαση του Συμβουλίου. Φαίνεται λοιπόν μια ενορχιστρωμένη ε, προσπάθεια να έχει αναπτυχθεί για να ανατραπεί το καθεστώς της Αλβανίας ως σοβαρού υποψηφίου. Δεν ξέρω γιατί. Μάλλον έχουν ξεκινήσει τα σοβαρά ήδη την προεκλογική τους εκστρατεία που πρόκειται να ολοκληρωθεί με την ε, προσφυγή στις κάλπες του χρόνου. Εγώ προσωπικώ θα ήθελα ο κόσμος, ο λαός της Αλβανίας να ε, λάβει το καθεστώς του υποψηφίου. δυστυχώ όμω η πολιτική τους οποίους έχουν επιλέξει φαίνεται να έχουν χαθεί σε μια περιδίνηση πολιτική. Και έτσι δεν θα μπορέσουν, μέχρι ότου κανονίσουν και αποφασίσουν τι προτεραιότητες θέλουν, δεν θα μπορέσουμε να του δώσουμε αυτό το καθεστώ. Και γι' αυτό παρακαλώ θερμά, κύριε Μπερίσα, κύριε Λάμα, για το καλό των πολιτών σα, για το καλό των λαών σα, του λαού σα, ελάτε πάλι στο δρόμο. Ευχαριστώ πολύ και τώρα ακούμε του λοιπού ομιλητέ, Ξεκινάμε με την κυρία Γιαννάκου για ένα μισή λεπτό. Πολύ κυρία Πρόεδρε σαφέστατα υποστηρίζουμε τη διάθεση και τις προσπάθειες της αλβανίας να γίνει μέλος της ευρωπαϊκής ένωσης και βέβαια συγχαίρω τον εισηγητή κύριο χουντή για την πάρα πολύ ισορροπημένη έκθεσή του. είναι φανερό βέβαια ότι το συμβούλιο θα κρίνει μάλλον ότι δεν πληρεί τις προϋποθέσεις η αλβανία δηλαδή δεν πληρεί κυρίως τα δώδεκα κριτήρια που έθεσε η ευρωπαϊκή επιτροπή για να μπορέσει η αλβανία να προχωρήσει και να αποκτήσει ευρωπαϊκή προοπτική ωστόσο αυτό μπορεί να αποτελέσει ένα έναυσμα για σταθερότερη πολιτική στην αλβανία για συνεννόηση μεταξύ των αλβανικών πολιτικών δυνάμεων και κυρίως για ρύθμιση ορισμένων θεμάτων που παραμένουν εκκρεμή όπως είναι η διαφθορά που υπάρχει ακόμα το οργανωμένο έγκλημα το ξέπλυμα χρημάτων καθώς και η διαφθορά στη δικαιοσύνη. επίσης στα θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων υπάρχουν προβλήματα κυρίως με τα ζητήματα της ιδιοκτησίας δεδομένου ότι υπάρχουν μειονότητες αναγνωρισμένες διεθνώς όπως η ελληνική μειονότητα. τέλος ε, κυρία πρόεδρε ε, σχολιάστηκε η στάση του κυρίου μπερίσα όταν εορτάζοντας τη βλόρα τα 100 χρόνια ε, της επετείου του κράτους που δημιουργήθηκε τότε για την αλβανία έκανε λόγο για πέντε χώρες στις οποίες βρίσκονται αλβανοί και αλβανικές μειονότητες. σήμερα επιχειρήθηκε η αλλαγή αυτού του σχολείου και έκανε τα πράγματα χειρότερα. λαμβάνοντας υπόψη ότι στη χώρα μας υπάρχουν μόνο αλβανοί οικονομικοί μετανάστες που εργάζονται και στέλνουν χρήματα στη χώρα τους και σε καμία περίπτωση δεν υπήρξε ποτέ αλβανική μειονότητα θα πρέπει να ξεκαθαριστεί προς την πλευρά αυτή ότι δεν είναι δυνατόν με μεγαλοειδιατισμούς και μια μυσαλλοδοξία να υποδέχονται τις ευρωπαϊκές αποφάσεις είναι προφανές ότι ο αλβανός πρωθυπουργός έκανε αυτή την κίνηση εθνικιστικού χαρακτήρα αναμένοντας την αρνητική για τη χώρα του απόφαση του συμβουλίου. πρέπει να του δοθεί ένα μήνυμα ότι η αλβανία δεν θα χάσει το παιχνίδι εκ των έξω αν συνεχίσει έτσι αλλά έχει μεγάλες πιθανότητες να το χάσει εκ των έσω. ευχαριστώ πολύ κυρία πρόεδρε. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει ο συνάδελφος Κύριλο για ένα λεπτό. Κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Θα ήθελα καταρχάς να αναφερθώ στην έκθεση και να ε, την επενέσω διότι περιγράφει πολύ ικανοποιητικά την κατάσταση της Αλβανίας και τις ε, συνθήκες που επικρατούν. Νομίζω ότι η Αλβανία έχει το δυναμικό για να ξεπεράσει τη δύσκολη κατάσταση που αντιμετωπίζει. Ωστόσο, θα πρέπει να εκφράσω και εγώ την ανησυχία μου σε σχέση με την εθνικιστική ε, ρητορία που διαχέεται. Μια ρητορία η οποία και με την επέτειο των 100 ετών από την ε, ίδρυση του κράτους επαναλαμβάνεται. Δυστυχώς, επί τη ευκαιρία λοιπόν αυτών των επαιτειακών εκδηλώσεων, ο Πρωθυπουργός της Αλβανίας μίλησε για τις περιοχές μεταξύ Ποτκόριτσα και Σκοπίων λέγοντας ότι ανήκουν στην Αλβανία. Τέτοιου είδους τοποθετήσεις μόνο σε, εθνο, σε ε, ε, διεθνικές εντάσεις μπορούν να οδηγήσουν. Πρέπει λοιπόν να αποσταλεί ένα σαφές μήνυμα προς την Αλβανία ότι τέτοιου είδους εθνικιστικές ρητορίες είναι αγαράδεκτες. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Το λόγο έχει ο κύριος Πόσελτ για 1,5 λεπτό. Κυρία Πρόεδρε. η Αλβανοί είναι ένας από τους αρχαιότερους κατά πάσα πιθανότητα λαούς της Ευρώπης και από το 1888 από το Κογκρέσο του Βερολίνου, από το Συνέδριο του Βερολίνου αναγνωρίστηκαν ως ανεξάρτητο κράτος. Ήταν ο μοναδικός λαός των Βαλκανίων ο οποίος δεν ε, ε, δεν έλαβε εκείνη την εποχή το καθεστώς ανεξαρτησίας και αναγνώριση ε, βρέθηκαν μέσα στη διελκυστίνδα μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων και μετά τις σφαγές στο Κοσφοπέδιο που περιγράφηκαν σε ένα πολύ εντυπωσιακό βιβλίο της εποχής εκείνης υπέστησαν μια γενοκτονία από την καταπίεση των Σέρβων της εποχής. Έτσι λοιπόν θα ήθελα να πω ότι σαφές είναι το εξής το να ε, εορτάζει κανείς ε, την εκατοντετηρίδα αυτών των γεγονότων και να μιλάει για ε, τους αδελφούς ανά τον κόσμο δεν είναι καταδικαστέο και αν δεν είναι πολύ ευφύης επιλογή πολιτικά. Οι Αλβανοί δεν ζητούν καμία αλλαγή συνόρων. Ούτε εμεί ζητούμε βεβαίω αλλαγή συνόρων. Θέλουμε να είναι εγγυημένα τα σύνορα και να είναι και προστατευμένα. Ωστόσο θα πρέπει να πούμε ότι έστω και αν δεν ήταν ευφυείς αυτές οι δηλώσεις, το να απαρνιόμαστε στους ε, Κωσοβάρους ε, την ε, ένταξη τους στην Ευρώπη, το να αρνιόμαστε για τους Αλβανούς τον της Σερβίας, ιδιαίτερα στην περιοχή του Πρέσοβο, ε, δικαιώματα και αναγνώριση μειονότητα, τότε προφανώ η κατάσταση θα επιδεινώνεται διαρκώ. Κάθε λαό έρχεται μια στιγμή όπου ε, αντιδρά στην καταπίεση. Και ναι, μπορεί να επικρίνουμε του Αλβανού, αλλά πρέπει να επικρίνουμε και του άλλου. Η Σερβία μέσα στο Σύνταγμά τη έχει ε, γράψει εδαφικέ διεκδικήσει ενάντια του πεδίου. και όμω έχει αναγνωρισμένο καθεστώ υποψηφίου για την ταξικράτου, όπω άλλωστε έχουν κάνει και άλλοι. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να δώσουμε μια ευρωπαϊκή προοπτική στην Αλβανία χωρί αλλαγέ συμφόρων και με προστασία μειονοτήτων για κάθε ε, μία από τις ε, μειονότητες των Αλβανών. Ευχαριστώ. Θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στον κύριο Τούσαφ που τη ζήτησε με τη διαδικασία ΚΑΤΣΙΑΕ. Παρακαλώ. Του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αξιολογούν την ενταξιακή πορεία της Αλβανίας με βάση τα κριτήρια των συνθηκών του μάστριχτ της κοπενχάγης της λισαβόνας της τέσσερις ελευθερίας του κεφαλαίου τη στρατηγική της ευρωπαϊκής ένωσης ευρώπη. 2020» καπιταλιστικές αναδιαρθρώσεις στην οικονομία για τη διείσδυση των ευρωπαϊκών μονοπωλίων στην αλβανία για την άγρια εκμετάλλευση των εργαζομένων των πλουτοπαραγωγικών πηγών πετρέλαιο φυσικό αέριο ρηκτός πλούτος και ταυτόχρονα ενίσχυση του αστικού πολιτικού συστήματος των κατασταλτικών μηχανισμών για τη χειραγώγηση του εργατικού κινήματος. τα εθνικιστικά και σοβινιστικά κηρύγματα και πολιτικές χρυσός κανόνας της αστικής τάξης αξιοποιούνται για την εκμετάλλευση των λαών στην ευρύτερη περιοχή των βαλκανίων. εκφράζουμε τη ριζική αντίθεση του κομμουνιστικού κόμματος της ελλάδας για την ένταξη της αλβανίας στην ευρωπαϊκή ένωση. οι λαοί αντιπαλεύουν την ενσωμάτωση νέων κρατών στην ευρωπαϊκή ένωση. οι πάλι για την αποδέσμευση από την ευρωπαϊκή ένωση είναι άρρηκτα συνεδεμένοι με την ανατροπή της εξουσίας των μονοπωλίων για τη λαϊκή εξουσία και οικονομία για την ανάπτυξη σχέσεων φιλίας και συνεργασίας των λαών στη βάση του αμοιβαίου ωφέλου. Ευχαριστώ κύριε Τούσα. Ο Επίτροπος Φούλα έχει τώρα εγώ. Μισό λεπτό κύριε Επίτροπε. Βλέπω μία μπλε κάρτα. Παρακαλώ. Είμαι απολύτως υπέρ της ένταξης της Αλβανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Τούσα ε, για το θέμα του καθεστώτος του υποψηφίου κράτους. Θέλω λοιπόν να ρωτήσω εάν μπορούν να αποφασίσουν μόνοι τους οι Αλβανοί αν θέλουν να προσχωρήσουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή αν θα πρέπει αυτό να είναι απόφαση των κομμουνιστών της Ελλάδας. ότι είναι κυρίαρχη η άποψη του λαού, του αλβανικού λαού, σε ό,τι αφορά την επιλογή που θα κάνει. Όμως όλοι ως πολιτικά κόμματα έχουμε ευθύνη να τοποθετηθούμε τόσο για την αλβανία όσο και για τις άλλες χώρες. για τους ίδιους όρους που ταχθήκαμε ενάντια στην ένταξη της ελλάδας στην ευρωπαϊκή ένωση ισχύουν οι ίδιοι όροι και λόγοι αυτούς που επικαλούμαστε και για την αλβανία. Ωραία. Το λόγο Ο Επίτροπος Φούλε. Uh, Κυρία Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη, είμαι ευγνώμων για την ευκαιρία που μου δίνεται να ανταλλάξουμε απόψεις για την ευρωπαϊκή προοπτική της ε, Αλβανίας. Το ψήφισμα αυτό στέλνει ένα σωστό μήνυμα στην Αλβανία. Αναγνωρίζουμε τις προσπάθειες που έχουν καταβάλει και, τους, ε, και και τα πολιτικά κόμματα και όλους τους ενδιαφερόμενους να εστιάσουν την προσοχή τους στην ε, διαδικασία μεταρρύθμισης. Όπως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έτσι και εμείς θεωρούμε ότι το μέλλον της Ασβανίας είναι κοντά σε αυτό της Ευρώπης και είμαστε διατεθειμένοι να δώσουμε καθεστώς υποψήφια προς ένταξη χώρας. Η Αλβανία όμως με τη σειρά της θα πρέπει να υποβάλει ε, ε, θα πρέπει να καταγράψει πρόοδο, κυρίως να γίνουν προσπάθειες στον τομέα του κανοδικαίου, του κράτους δικαίου. Θα πρέπει να υιοθετήσει μια ισχυρή, αξιόπιστη πολιτική, η οποία θα αποβεί υπέρ των όλων των πολιτών της Αλβανίας. Ευχαριστώ πολύ. Commissario, la parola al Ministro Κυρία Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη, κύριε Επίτροπε, η ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να προκύψει μόνο μετά από σημαντικές προσπάθειες σε εθνικό επίπεδο αλλά και σε επίπεδο συλλογικής δέσμευσης. Η Αλβανία χρειάζεται να εξασφαλίσει έναν ε, σταθερό και επικοδομητικό πολιτικό διάλογο. Η υποστήριξη από πλευρά των Αλβανών πολιτών στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση αποτελεί μια σημαντική βάση πάνω στην οποία οι πολιτικοί ηγέτες μπορούν να ανεκοδορήσουν μια κοινή πλατφόρμα προς το συμφέρον της χώρας στο σύνολό της. Θα ήθελα να τελειώσω τονίζοντας ε, τη σημαντική πρόοδο που έχει επιτευχθεί στην Αλβανία την προηγούμενη χρονιά απέδειξε, έδειξε ότι διαθέτει πολιτική βούληση, κατέληξε σε αυτά αποτελέσματα και κατάφερε να εφαρμόσει μεταρρυθμίσεις. Έχω την απόλυτη υπεποίθηση ότι το υψηλό επίπεδο δέσμευσης θα έχει συνεχιστεί και ότι στο μέλλον θα δούμε περαιτέρω θετικές εξελίξεις κατά τη διάρκεια του 2013. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ έλαβα μία πρόταση ψηφίσματος στο πέρα συζήτηση. Πέρα συζήτηση, ψηφοφορία αύριο στις 12. Ώρα... Περνάμε